Παρακαλώ, καθίστε. Για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη συνεδρία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την βιωσιμότητα και σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών. Θα έχετε δύο λεπτά ο καθένας αυτό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό όσων θα ζητήσουν το λόγο. Υπάρχουν και αιτήματα ε, υποβολής ερωτημάτων από, από το πρώτο μέρος της συνεδρίας δεν θα τα ακούσουμε γιατί το αντικείμενο της ε, συζήτησης ε, τώρα είναι διαφορετικό. Εάν κάποιος ζήτησε το λόγο ε, την προηγούμενη φορά στο πρώτο μέρος της συνεδρίας και δεν του δόθηκε, πρέπει να τον ξαναζητήσει τώρα το λόγο για το θέμα που μας απασχολεί. Και αν δω ότι δεν σας δόθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίας, θα σας δώσω προτεραιότητα. Εάν όμως θέλετε το λόγο, πρέπει να τον ξαναζητήσετε. Έχουμε δύο εισηγητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την διάδα των μέτρων που είναι η συνέχεια της εξάδας των μέτρων. Ε, το two-pack ως συνέχεια του six-pack δηλαδή. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους εισηγητές εκ μέρους των κοινοβουλίων τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Οικονομικών από το Κοινοβούλιο της Λετωνίας και μετά τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων ε, του Αυστριακού Συμβουλίου του κυρίου, τον κύριο Κρέινερ, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε ερωτήσεις από τους παριστάμενους. Λοιπόν, να υποβάλλετε νέες κάρτες με, στις, τις οποίες θα έχετε συμπληρώσει αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο και αν το κάνατε στην πρώτη συνεδρία και δεν σας δόθηκε, αυτό θα το προσέξω ιδιαίτερος. Ευχαριστώ. Ε, ο πρώτο συζητήτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι ο τρόπος με τον οποίο ο Άλλα Λαμασίου παρουσίασε αυτή τη συνεδρία λέγοντας ότι από τη μία θα πρέπει να καθίσουν οι υπέρμαχοι της ε, ε, λιτότητας ήταν κάτι το οποίο ε, είχε αρνητικό αντίκτυπο στους παριστάμενους. Ωστόσο, θα ήθελα να παρουσιάσω αυτή την διάδα μέτρων τα οποία συμπληρώνουν την εξάδα μέτρων που προηγήθηκε. Είμαι εισηγητής ε, σε ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία και εποπτεία του προπολογισμού των κρατών μελών, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ως προς τη δημοσιονομική σταθερότητα και είναι ήδη ε, μέλη της ζώνης του ευρώ. Και είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ε, οικονομικής κρίσης, της κρίσης εθνικού χρέους, την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το κείμενο αυτό προσπαθούμε να αντλήσουμε τα διδάγματα της κρίσης και να υποβάλουμε συγκεκριμένα προτάσεις. Και μάλιστα ε, να μιλήσουμε για τις συνέπειες της υπερχρέωσης των κρατών. Δεν χρειάζεται να σας δώσω λεπτοπο, λεπτομέρειες επ' αυτού, διότι η υπερχρέωση των κρατών μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες ως προς την κατάσταση του εν λόγω κράτους, αλλά και ως προς την κατάσταση την εργασιακή, την οικονομική και την κατάσταση ως προς τους δείκτες απασχόλησης στο ίδιο αυτό κράτος, αλλά και στα υπόλοιπα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η εξάδα των μέτρων για να ενισχυθεί η σταθερότητα και η οικονομική μεγέθυνση στους ε, κόλπου της ζώνης του ευρώ. Το, η εμπειρία μας διδάσκει ότι ορισμένα κράτη-μέλη υποχρεώθηκαν να ζητήσουν δημοσιονομική συνδρομή, χρηματοδοτική συνδρομή. Και βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε απαραίτητα εργαλεία και όργανα όταν ζήτησαν αυτή την χρηματοδοτική ε, συνδρομή και ε, Γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δύο κείμενα τα οποία συζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον όσον αφορά στο πρώτο κείμενο, δεν ε, απαιτεί μεγάλες τροποποιήσεις. Θα ήθελα να πω ότι, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ κατά, το τελευταίο, κατά τη τελευταία του συνεδρίαση τοποθετήθηκε επί αυτής της έκθεσης χωρίς να ε, παρουσιάσει σημαντικές τροποποιήσεις και τροπολογίες επί των προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διάφορες προσθήκες και προβληματισμοί θα ενσωματωθούν στο κείμενο. Ως προς τις προσθήκες, για να διευκρινιστεί καλύτερα η νομική κατάσταση ε, την οποία δημιουργεί η διακυβερνητική συνθήκη. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε στο κείμενο του κανονισμού να επανεισαχθούν οι διατάξεις στις συνθήκες που μπορούν να επανεισαχθούν. Δηλαδή, πολλές από αυτές τις διατάξεις εκτός από το χρυσό κανόνα, ο οποίος κατά την άποψή μου ε, άπτεται αμυγός στις συνθήκες αυτής της διακυβερνητικής και ε, ουσιαστικά έγκυται στο εταιρικό δίκαιο, δηλαδή είναι ένα σύμφωνο μεταξύ μετόχων ουσιαστικά. Άρα, Στόχος είναι στο κείμενο και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται κάποιες από τις τροπολογίες μου να ενταχθούν σε αυτό το κείμενο οι διατάξεις της διακυβερνητικής συνθήκης που δεν έχουν ακόμα επικυρωθεί. Θεωρούμε ότι το Συμβούλιο και περιέργως το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ δεν ζήτησε ε, ε, το Συμβούλιο να έχει λόγο επί των προτάσεων που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το θέμα αυτό της ενισχυμένης εποπτείας. Και μου φαίνεται μάλιστα αρκετά περίεργο το γεγονός ότι το αρχικό κείμενο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο Συμβούλιο και μου φαίνεται απολύτως περίεργο το Συμβούλιο το ίδιο να μην ζητεί να περιληφθεί αναφορά στον εαυτό του. Και αν το έκαναν εσκεμένα θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε το γιατί δεν ζήτησαν να ε, συμπεριληφθεί αναφορά στους εαυτούς τους, στο Συμβούλιο δηλαδή. Ε, τέλος, θα ήθελα επίσης να πω και το εξής κάτι το οποίο γνωρίζει η διάσκεψη των Προέδρων και μάλιστα ε, είναι θετικά διακείμενη. Καλό θα ήταν να αντλήσουμε τα διδάγματα ε, από την εξής κατάσταση που έχουμε διαπιστώσει σήμερα. Ε, τα κράτη που βρίσκονται στο όριο της κήρυξης τάσης πληρωμών δεν μπορούν να υποστηρίζουν να αντέξουν την πίεση που υφίστανται αν δεν ληφθούν ε, επιπρόσθετα και συμπληρωματικά μέτρα. Προτείνουμε λοιπόν ε, και για τα κράτη να ισχύσει αυτό ένα σύστημα νομικής προτεστασίας που ισχύει και για τις, για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το κράτος να έχει στη διάθεσή του ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανακάμψει, προκειμένου να συνέλθει, προκειμένου να ε, εφαρμόσει αυτά τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης είναι ένα θέμα επί του οποίου θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και σίγουρα θα δώσει λαβή για πολύ μεγάλες συζητήσεις γιατί βασικό πρόβλημα θα είναι η διατύπωση ενός τέτοιου είδους μηχανισμού και πώς αυτή ε, θα συνδυαστεί με τις δημοκρατικές αρχές που μας διέπουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ελίσα Φερέιρα. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως μόλις είπε ο συνάδελφος Γκοζές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε παράγοντα κλειδί στις διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα για το εξαπλό πακέτο που τέθησε ισχύ το Δεκέμβριο, 13 Δεκεμβρίου και βρισκόμασταν ακόμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης και δημοσίευσης του εξαπλού πακέτου, δημοσίευση που έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2011 και στην ίδια ημερομηνία η Κομισιόν δημοσίευσε δύο νέες προτάσεις κανονισμού για να εντατικοποιήσει την ε, παρακολούθηση και υποπτία των κρατών μελών που αποτελούν μέρος ε, του Ευρωζώνης. Για τα δύο αυτά επιπλέον κείμενα εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ενώ εντωμεταξύ η διακυβερνητική συνθήκη, η δημοσιονομική, ε, ή μάλλον η... Το εταιρικό σύμφωνο, όπως το πεκάλεσε ο συνάδελφος, το Fiscal Compact, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. από τους στόχους μας ε, για αυτή τη δουλειά είναι να δώσουμε μια συνοχή στα όσα γίνονται και ιδιαιτέρως να μετατραπεί αυτό το διπλό πακέτο σε κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο. Ο συνάδελφος Γκοζές εργάζεται για τις εκθέσεις αυτές. Εγώ εργάζομαι για την πρωτοβουλία της Κομισιόν που είναι γνωστή ως 421 για το συντονισμό των δημοσιονομικών προτάσεων. Και εκεί η Κομισιόν έχει επιπλέον εξουσίες να ζητήσει δηλαδή ενημέρωση, να κάνει έλεγχο και να αξιολογήσει τον κίνδυνο μη πλήρωσης των δημοσιονομικών στόχων των χωρών. Ε, αυτή τη στιγμή οι προτάσεις μου έχουν ε, τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτον, είναι σημαντικό να υπάρχει μια προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τις ε, διαδικασίες, τις ε, ε, εθνικές νομοθετικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό να μην ε, απολεστεί η εθνική ευθύνη και η δυνατότητα διαφάνειας και η δυνατότητα να αποδίδεται ο παράγοντας της δημοκρατικής νομιμότητας στη δημοσιονομική διαδικασία και γι' αυτό οι προθεσμίες που αυτή τη στιγμή προβλέπονται στην πρόταση της Κομισιόν πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος ε, στην εθνική νομοθετική διαδικασία να εξελίσσεται με κάθε κάθε κανονικότητα, με κανονικό ρυθμό και με την άσκηση της δημοκρατίας και της εθνικής ιδιοποίησης του κανονισμού που απαιτείται από τη δημοκρατία. Αυτό είναι ένας από τους ε, πρώτους στόχους. Ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με την ισορροπία ανάμεσα στις εξουσίες της Επιτροπής που θέλει να ενισχύσει αυτό το κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά τον στόχο εγγύησης της εθνικής νομιμότητας για το μέλλον και την εξέλιξη της κάθε χώρας μέλους, αλλά ταυτόχρονα το ρόλο που θα πρέπει να εγγυόμεθα στο Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις μεμονωμένες χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από την άλλη πλευρά τα διάφορα άλλα όργανα, δηλαδή Συμβούλιο, Κομισιόν, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος. Ένας τέταρτος στόχος είναι να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην ετήσια δημοσιονομική διαδικασία και τις συστάσεις και νομοθετικά κείμενα που εκπονούνται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δηλαδή σε εθνικό επίπεδο την ανάγκη ε, να ε, υπάρξουν εθνικά προγράμματα ε, μεταρρύθμισης, σταθερότητας και ανάκαμψης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την οικονομική ανάκαμψη και την αξιολόγησή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γενικές εργασίες για την απασχόληση, αλλά και έχουμε και τα αποτελέσματα για την μακροοικονομική ανισορροπία η ανάλυση από πλευρά της Κομισιόν των όσων είναι η δημοσιονομική χρήση κάθε χώρας θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την δημοσιονομική ισορροπία σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλησης και διόρθωσης των ενδεχόμενων ανισορροπιών σε επίπεδο δημοσιονομικού, αλλά αυτή η αυτό το εγχείρημα να είναι απόλυτα συμβατό με τις συστάσεις τις αιτήσει αλλά και τις πολιετήσεις για κάθε χώρα. Τέλος, αυτή τη στιγμή είμαι πεπισμένη και ήδη αυτό έχει παρουσιαστεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Ο επόμενος στόχος είναι αυτό το μεγάλο εγχείρημα για μεγαλύτερο έλεγχο για την ε, οικονομική ισορροπία και τη δημοσιονομική ισορροπία των χωρών να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα συντονισμού όσον αφορά τη διαχείριση του κρατικού χρέους και να υπάρχει δέσμευση για δυνατότητα πρόσβασης στη συγκεκριμένη πορεία αντιμετώπισης του κρατικού χρέους, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει επιχείρηση διάσωσης από το Ταμείο Διάσωσης για τις ε, χώρες που δεν καταφέρουν να κλείσουν το έλλειμμα. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ως Κοινοβούλιο ότι προς εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, next... Ευχαριστώ και εγώ. Ας ακολουθήσει ο κύριος Ρίας από την Λετωνία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Δημοσιονομική εξυγίανση που να στηρίζει την ανάπτυξη. Υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πολλοί φοβούνται ότι οι στόχοι αυτοί είναι αντιφατικοί. Ίσως όμως έχει έρθει ο χρόνος που μας καθιστά απαραίτητο να προσπαθήσουμε να συμβάσουμε τα δύο αυτά αντιφατικά ε, στοιχεία. Είναι απαραίτητο να εξηγερθούν τα δημοσιονομικά αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα από όλα, δηλαδή την υπέρβαση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη και να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στις διάφορες μέλη και βέβαια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικότερα. Βιώσιμες λοιπόν μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί η ανεργία, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη που ούτως ή άλλως αποτελούν σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξε καμία ουσιώδης βελτίωση στους τομείς αυτούς. Νομίζω όλοι λίγο πολύ θα συμφωνήσετε ότι για ότι να επιτευχθεί η ε, δημοσιονομική εξυγένση είναι στην πραγματικότητα σήμερα πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια, δηλαδή πρώτα να, συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουν όλοι δηλαδή σχετικά με τους στόχους, δεύτερον να γίνει με συνέπεια η μεταρρύθμιση και τρίτο και πιο σημαντικό, να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις με κοινωνική αποδοχή. Αυτά τα τρία πράγματα βέβαια πρέπει να αλληλοσυνδέονται και η αλληλοσύνδεση αυτή δεν μπορεί να λησμονείται. Εφόσον επιτευχθούν αυτά μπορεί να επιτύχει κανείς ε, και παραπέρα. Κάτι καταφέραμε στη Λετωνία. Μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε μια υπερθέρμανση της οικονομίας και μπορέσαμε να υπερβούμε την κρίση με την καθοδήγηση της κυβέρνησης του Βάλτης τον Πρόσκης, μπορέσαμε να μειώσουμε σημαντικά το δημοσιονομικό μας έλλειμμα, να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας κατά 5,3% στο 2011. Η στρατηγική που επέλεξε η Λετωνία για να ξεπεράσει την κρίση οδήγησε και σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή που προβλεπόταν αρχικά. Και μάλιστα και το δημοσιονομικό μας έλλειμμα μειώθηκε από τα 6% που προβλεπόταν στα 4%. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση που να είναι φιλική προς την ανάπτυξη. Βέβαια, μια ιστορία επιτυχίας όπως η δική μας ίσως να μην μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες ε, χώρες. Η λύσεις ωστόσο που επιλέξαμε εμείς ίσως είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και αλλού. Το νομοθετικό πακέτο, το λεγόμενο six pack, η δέσμη των 6 μέτρων, εγκρίθηκε το προηγούμενο φθινόπωρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σημαντικές προτάσεις πρωτοβουλειών και βάσει, στη βάση αυτών δημιουργήθηκε και η νέα δημοσιονομική συμφωνία. Αυτά είναι σημαντικά για να ομαλοποιηθεί η δημοσιονομική κατάσταση και στο μέλλον θα επιτρέψουν και την αποφυγή κρίσεων. Φέτος η Λετωνία συνεργάστηκε και ε, επέτυχε σημαντικές πρόοδους και στη συνεργασία της με το, με το, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε υποβάλει τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα είναι σύμφωνες και με τη νέα δημοσιονομική συνθήκη με πρώτα τροπολογίες στον προϋπολογισμό μας και στην οικονομική διαχείριση, οικονομική διακυβέρνηση και τη σχετική νομοθεσία που προβλέπουν νέα διαδικασία για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού με ειδική νομοθεσία κάθε ε, χρόνο η οποία θα θεσπίζει τα ανώτατα όρια των δαπανών σε αιτήσια βάση. Επίσης, σχεδιάζονται τροπολογίες σε νομοσχέδια που θα βάζουν τις, βάση, βάσεις για έναν προϋπολογισμό υπό Δεύτερο, η νομοθετική εργασία έχει αρχίσει για τροποποίηση του συντάγματος που θα περιλάβουν διατάξεις για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με την έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, επεξεργαζόμαστε νομοσχέδιο δημοσιονομικής λιτότητας που θα προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις για την ετήσια διαχείριση του προϋπολογισμού. Ήδη το νομοσχέδιο αυτό έχει εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση, προβλέπει τις προϋποθέσεις για εξυγίανση του προϋπολογισμού και εκτός αυτού λάβαμε και την απόφαση πριν εγκρίνουμε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού να ελέγχουμε την συμμόρφωσή του με την Δημοσιονομική Συμφωνία. Πιστεύουμε ότι μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους θα έχει συμμορφωθεί πλήρως η λετωνική νομοθεσία με την Δημοσιονομική Συμφωνία. Πιστεύω ότι όλες οι Εθνικές Βουλές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις λήψεις αποφάσεων για την δημιουργία μιας Ευρώπης δημοσιονομικά εξηγιασμένης και με βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω η σύντομη αυτή παρέμβασή μου να σας κάνει να πιστέψετε ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η κρίση με τα μέτρα αυτά. Ε, η Πρόεδρος, υπενθυμίζω, έχω, ε, ακόμη έχω πέντε εγγεγραμμένους ομιλητές. Ίσως δεν έχουμε τόση μεγάλη πίεση χρόνου. Εάν θέλετε ωστόσο να μιλήσετε, στείλτε μας μια κάρτα ακόμη. Ο κύριος Κράμερ του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς οι βουλευτές κάναμε σκληρή προσπάθεια για να δώσουμε απαντήσεις στην οικονομική κρίση που έπληξε τον κόσμο και την Ευρώπη βέβαια μετά το 2008. Η δημοσιονομική κρίση που έγινε και η οικονομική κρίση σε όλες τις χώρες μας και σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης οδήγησε εν τέλει και σε κοινωνική κρίση με πάρα πολύ υψηλή ανεργία και κυρίως που πλήττει τους νέους καθώς επίσης και ε, με σοβαρότατα δημόσια ελλείμματα. Οι βασικές αιτίες της οικονομικής κρίσης είναι πρώτα οι μη ρυθμισμένες οικονομικές αγορές, οι ελλείψεις ισορροπιών μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης και τρίτο η άνηση κατανομή του πλούτου και του εισοδήματο μέσα στις κοινωνίες μας. Πρώτα για τις μη ρυθμισμένες οικονομικές αγορές. Νομίζω ότι εκεί πήραμε πολλά και σημαντικά μέτρα για να θεσπίσουμε καλύτερη ρύθμιση, καλύτερες διατάξεις από ότι πριν από την κρίση υπάρχουν ορισμένες ακόμα που έρχονται στον αγωγό όπως λέμε, ωστόσο ένα σημαντικό βήμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και εννοώ τον ε, φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοπιστωτικές αγορές θα συμβάλλουν στο κόστος αντιμετώπισης της κρίσης που επέφεραν οι τέλη στις κοινωνίες μας. Το δεύτερο για τις ελλείψεις οροπιών μεταξύ των οικονομιών μας. Νομίζω ότι με το 6 pack και το 2 pack το ευρωπαϊκό εξάμενο και ούτε καθεξής έχουν όντως ληφθεί σημαντικά μέτρα για να αυξηθεί η διαφάνεια ε, στη σχέση μεταξύ των χωρών μας, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας, αλλά και να ενισχυθεί και η εποπτεία. Τα μέτρα αυτά ωστόσο θα έχουν νόημα μόνο εάν εν τέλει χρησιμοποιήσουμε όντως αυτά τα μέτρα που προσφέρουν αυξημένη διαφάνεια και εποπτεία για να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε και θα αναχρηματοδοτήσουμε τις χώρες μας. Είτε με ομόλογα έργων, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης. Αυτό είναι λιγότερο σημαντικό. Αυτό που χρειαζόμαστε ωστόσο είναι χαμηλότερα επιτόκια, ανεξαρτησία από τις οικονομικές αγορές για τη χρηματοδότηση των χωρών μας. Και το τρίτο στοιχείο είναι η άνηση κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Εκεί νομίζω έχουμε πράξει τα ελάχιστα. Το κενό, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων μεγαλώνει διαρκώς. Εξακολουθούμε να επιβαρύνουμε φορολογικά την εργασία και πολύ περισσότερο από ό,τι επιβαρύνουμε το κεφάλαιο και την αξία ή την υπεραξία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό το 1% της κοινωνίας μας που είναι οι πλούσιοι να πληρώσουν και αυτοί δίκαιο και ίσο μερίδιο. Αυτό πρέπει, αυτή την προσπάθεια πρέπει να την επιταχύνουμε. Και αν εξετάσουμε την τελευταία σημαντική οικονομική κρίση και πώς οι Ηνωμένε Πολιτείε την ξεπέρασαν, είναι ότι βάλαν αυτό το 1% να πληρώσει και αυτό δίκαιο μερίδιο. Ο Φρανκ Ρούσβελτ τότε και οι πρόεδροι που τον διαδέχτηκαν στερέωσαν Έβαλαν βέβαια μέχρι και 70% φορολογία, ίσως είναι υπερβολικό αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει λόγος και υπάρχει και χώρος για να μειωθεί αυτή η ανισότητα. Εν συνόψη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μένουν ωστόσο πολλά να γίνουν ακόμη. Τα τέσσερα που έχω να πω είναι εξή. Πρώτον, ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεύτερο, ανεξαρτησία από τις χρηματοπιστωτικές αγορές τρίτο το 1% να πληρώσει το δίκαιο μερίδιό του και το τέταρτο η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με αύξηση της εργασίας, με αύξηση της απασχόλησης και όχι με παραπέρα λιτότητα. Αυτά τα κάνουμε και στην Αυστρία βέβαια, αλλά είναι το ίδιο σημαντικό να υπάρξει ανάπτυξη σε όλες τις χώρες μας. Όχι αύξηση της ανεργίας, αλλά μείωση της ανεργίας. Τα λέω αυτά και προερχόμενο από μια χώρα η οποία χαίρει ευτυχώ σχετικά χαμηλών επιπέδων ανεργία, Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί και είναι πρόβλημα. Επιτρέψτε μου ακόμη να σχολιάσω μια συνέντευξη ενό υψηλού αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έδωσε στο Wall Street Journal πριν από λίγε μέρε και που είπε ότι χάθηκε πλέον το κοινωνικό ε, μοντέλο της Ευρώπης. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αντίθετα, στις χώρες εκείνες όπου έχουμε ισχυρά συστήματα κοινωνικής ευημερίας, αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν καλύτερα, ευκολότερα την κρίση από εκείνες που δεν τα έχουν. Δεύτερο είναι ότι ποτέ δεν είδα εγώ τις επερχόμενες εκλογές ως ρίσκο ή ως πρόβλημα. Αντίθετα, θα θεωρούσα το να μην επίκυνται εκλογές ότι είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαι δημοκράτης. Και το τρίτο είναι ότι το πρώτο που διαβάζω το πρωί δεν είναι τα stock markets, είναι το ποσοστό της ανεργίας. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much. Everybody, we can now move. Ευχαριστώ. Περνούμε τώρα στις συνεισφορές των παριστάμενων μόνο από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ζητήσει το λόγο και αυτό είναι εξαιρετικό για να μπορέσουν να δουλέψουν οι εισηγητές μας. Διπλάσιοι τελικά έχουν ζητήσει το λόγο από ό,τι στην αρχή. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αν θέλετε άλλοι το λόγο παρακαλώ να τον ζητήσετε. Φιλίπ Μαρτίνη από την Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση στην κυρία Φερέιρα, η οποία στην παρέμβασή της μίλησε για ένα ταμείο για το εθνικό χρέος χωρών οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ακόμα δυσκολίες. Πώς συνδέεται αυτό με τον υφιστάμενο μηχανισμό ή με τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε. Από εκεί και πέρα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επιμείνω στη σημασία που έχει κατά την άποψή μου ε, να υπάρχουν σχέδια ε, προϋπολογιστικά δηλαδή σχέδια προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά που θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου και παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού ε, μεσοπρόθεσμη το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου. Ως προς τα αιτήσια σχέδια προϋπολογισμού. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η διαδικασία μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις και δεν θα πρέπει αυτό να μας, να μας σοκάρει. Ε, άμεσες επιπτώσεις στην εθνική νομοθετική διαδικασία. Η κυβέρνηση που Υποβάλλει προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο στη Σύνοδο του Οκτωβρίου θα πρέπει να τον τροποποιήσει τελικά ε, πριν από το τέλος ε, της συζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί κάτι. Οι ενδείξεις που θα πρέπει να δίδονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, διαμορφώνουν μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς τους στόχους ε, βάσει των οποίων θα εξελιχθούν οι δαπάνες και ως προς ε, τις προϋποθέσεις για να λάβουν χώρα οι δαπάνες αυτές. Δηλαδή, εάν ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένος κανόνας, μία συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει το κράτος μέλος να είναι σε θέση να εξηγήσει και να τεκμηριώσει τις δαπάνες αυτές αναδημοσιονομική γραμμή. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Στη Γαλλία έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εξετάζουμε δύο σχέδια. Ένα σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους και ένα νόμο για την χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και είναι και ο αρμόδιος συνάδελφος εδώ για να το σχολιάσει. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, ε, κάτι το ξεχωριστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν αυτό να το ταιριάξουμε με τα πηγενέλα που αναγκαστικά θα γίνονται ε, στο πλαίσιο αυτού του σχέδιου προϋπολογισμού. Θα ενοποιήσει τα δύο έγγραφα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έσοδα πιο συγκεκριμένα. Ε, θα ήταν χρήσιμο να εμβαθύνουμε ως προς αυτό το θέμα. Αυτό καταρχάς, κατά δεύτερο λόγο, ως προς τον δημοσιονομικό προγραμματισμό Ένα σημείο του κειμένου το οποίο δεν κατανόησα πολύ καλά είναι η διαφορά μεταξύ των μεσοπρόθεσμων σχεδίων προϋπολογισμού από τη μία και των προγραμμάτων σταθερότητας έτσι όπως έχουν καταρτιστεί μέχρι σήμερα από την άλλη. Τα πρώτα αντικαθίστανται από τα δεύτερα. Ε, ποιες είναι οι μεθοδολογικές ε, διαφορές ε, μεταξύ των δύο εγγράφων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήταν χρήσιμο, εκτός από ερωτήσεις, αν έχετε και προτάσεις να τις υποβάλλετε, αλλά στο τέλος ε, να έχουμε πρώτα τις ερωτήσεις. Να δώσω το λόγο στον κύριο Χάρισον, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή των Λόρδων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εγώ είμαι μέλος της αντιπολίτευσης, όπως όμως είπε και ο Ντέιβιτ Λίτινγκτον, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, ε, καλωσορίζεται στη Βρετανία η έννοια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής ε, ΙΜΑΚ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τότε μιλούσαμε για τις ευρείες οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι αναβάθμιση, ένα παράδειγμα αναβάθμισης του παλαιότερου εγχειρήματος. Τον περασμένο Μάρτιο δημοσιεύσαμε την πρώτη μας έκθεση για την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και ε, θεωρήσαμε ότι η βασική αιτία ήταν έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας και δεν ήταν καλό, δεν είναι ωραίο να κλωτσάει κανείς μια χώρα όταν βρίσκεται εξαπλωμένη στο έδαφος. Και μάλιστα αυτά υπήρχαν και στην έκθεση την ε, διάδοχη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα και ήσασταν εσείς μάρτυρες. Και είπαμε ότι στην έκθεση αυτή ότι ε, δόθηκε προτεραιότητα στη λιτότητα. Καλό θα ήταν ο πρόεδρος Μπαρόζο όταν αναφέρεται στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς να είναι προσεκτικός. Νομίζω ότι αν είχαμε πραγματικά ενιαία αγορά δεν θα είχαμε μπει, δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δανείζει ουσιαστικά τις τράπεζες, αυτό είναι βοηθητικό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεφεύγει από τα όρια τα οποία ορίζονται στο καταστατικό της, γιατί ακολουθεί αυτή την πολιτική του quantitative easing, αλλά δεν επαρκεί. Ως προς το ευρωομόλογο, ε, δεν έγινε λόγος γι' αυτό από τον πρόεδρο Μπαρόζο. Ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε για ομόλογα έργων, project bonds. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Οι συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα ήταν πολύ σημαντικές για την αναζωπήρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καλωσορίζουμε στην ε, έκθεσή μας αυτή την τριάδα των μέτρων, το πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα, Τώρα δεν έχει σημασία να απαιτείται ένα, τρει ή δύο, τρει ή πενήντα δις ευρώ για να ανακεφαλοποιηθούν και να εξηγιαθούν οι τράπεζες. Εμείς ως Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσαμε να μην υπογράψουμε, να μην προσχωρήσουμε σε αυτή την συνθήκη και έτσι η Βουλή των Λόρδων θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος οι υπόλοιπε ε, χώρε μέλη να μην προχωρήσουν. Και η Βουλή του Δόδων θεωρεί επίσης ότι η ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς απειλείται και ε, θα ήταν περισσότερο προστατευμένοι εάν και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούσε στη συνθήκη αυτή. Εμείς στη Βουλή των Λόρτων είμαστε υπέρ λοιπόν της υπογραφής. Ε, θα προστατευτεί περισσότερο η ενία αγορά, θα ε, δρομολογηθούν τα θέματα των υπηρεσιών και του φόρου επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντική τρόποι αύξηση των εσόδων. Καλό θα ήταν ο πρόεδρο Παρόσο να μα είχε πει γιατί ήταν κατά όλων αυτών ε, μετά από συμβουλέ από το οικονομικό του επιτελείο και από το επιτελείο που είχε να κάνει με τον προπολογισμό. Και γιατί ε, μετριάστηκε η πρόταση του φόρου ε, επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Από ό,τι κατάλαβα, είναι ανοιχτή στις προτάσεις και ίσως θα έπρεπε να αντιγραφεί ε, αυτή η ιδέα των τελών χαρτοσύμου που έχουμε εμεί στη χώρα μου. Τώρα, ως προς τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, θα ήταν κακή ιδέα να υπάρξει ευρωπαϊκή ειδικό Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, ο οποίος να είναι το ε, τέκνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι να έχουμε ένα πλαίσιο για προϋπολογισμό. Το σημαντικό είναι όμως ο προϋπολογισμός να κινητοποιεί την Ευρώπη, να έχει ευελιξία, έτσι ώστε η το όραμα για την Ευρώπη του 2020 δεν οδηγήσει ε, σε υπονοόμευση του Ταμείου Συνοχής. Καλό θα ήταν να δοθεί καλύτερος ορισμός της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Να γνωρίσουμε δηλαδή γιατί πρέπει να γίνονται πράγματα επιπρόσθετα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Αν όλοι μιλήσουν τόσο πολύ όσο εσεί, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσει. Αυτό είναι το δίλημα, βεβαίω, που αντιμετωπίζω εγώ ω Πρόεδρο. Να ακούσουμε τη συνάδελφο από την τον συνάδελφο από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου Λαμασούρου στο τέλος του προηγούμενης συνόδου στην οποία είχα εγώ ενταχθεί ήθελα να πω ότι θα θέλαμε εδώ να διευρυνθεί ο διάλογος ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις Επιτροπές προπολογισμού Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο στην εξέταση του εξαπλού πακέτου μαζί με την εισηγήτρια την κυρία Φερέιρα και τον Τζιόγκο Φέιο ε, και τώρα επεξετάζουμε το διπλό πακέτο αλλά βλέποντας την, από την προοπτική μιας χώρας όπου υπάρχει μεγάλη συνένεση κοινωνική και πολιτική γύρω από το πρόγραμμα μεταρρύθμισης που έχει διαπραγματευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση και βλέποντας από μια πορτογαλική προοπτική θεωρούμε, βλέπουμε μάλλον ότι είναι το πιο απαραίτητο σε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συνεδριάσεις, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να συμβάλλει ώστε να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη και Ευρώπη ε, εγκαίρος, έτσι ώστε να είναι προφανές ότι το πρόβλημα που έχουμε είναι πρόβλημα ε, ε, σφαιρικής απάντησης από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ιταλικό, ισπανικό, ιρλανδικό, πορτογαλικό ή ελληνικό το πρόβλημα μόνο. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί περισσότερο συντονισμό και λιγότερο εθνικισμό, που απαιτεί περισσότερη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών, συντονισμό, περισσότερη ελληνική και λιγότερη, λιγότερο απομονωτισμό και ε, υπεροχή των εθνικών προοπτικών. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτήν την ε, συνθήκη τη δημοσιονομική, βλέποντας το εξαπλό και το διπλό πακέτο. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δίνεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στο, στις πτυχές μάλλον δημοσιονομικού συντονισμού. Δεν γίνεται αντίστοιχη όμως προσπάθεια για συντονισμό των ε, ε, φορολογικών πολιτικών, ας πούμε, ώστε να μην συμβεί όπως στην Πορτογαλία που ένα μεγάλο μέρος των εταιριών που ήταν στο χρηματιστήριο για φορολογικούς λόγους μεταφέρθηκαν σε φορολογικού, τις έδρες τους μετέφεραν σε φορολογικούς παραδείσους εντός της Ένωσης. Δεν γίνεται αντίστοιχη υπάρχει προσπάθεια ούτε για το συντονισμό των πολιτικών πρόθεση τη ανάπτυξη. Δεν γίνεται ε, εντάξει, ισότιμη μάλλον προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων της ανεργίας. Ούτε προσπάθεια αντίστοιχη γίνεται για την ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ε, βλέπουμε ότι δεν γίνεται κανένα, καμία συντονισμένη παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο, από ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε για τη δημιουργία ε, για αυτού του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των ευρωομολόγων, ούτε σε αυτό που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής στα ομόλογα έργου. Δεν γίνονται αρκετές προσπάθειες και γι' αυτό το εξάμεινο έχει νόημα αν ο οικονομικός συντονισμός σήμαινε περισσότερη Ευρώπη και επιστροφή στο ευρωπαϊκό πνεύμα και όχι σε μια ιδέα διχόνοιας ε, ε, μιας Ευρώπης όπου κυρίως οι μεγαλύτεροι ξεκινούν παραβιάζοντας το σύμφωνο σταθερότητας ενώ παριστάνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι όλων αλλά μόνο κάποιων και παρά την εθνική προσπάθεια που καταβάλουν όλες οι χώρες μας και όπου η Πορτογαλία με μια πολύ έντονη εσωτερική συζήτηση ε, προσπαθεί να συνδυάσει τη λιτότητα με την ανάγκη ανάπτυξης και πολιτικών υπέρ της απασχόλησης. Μια προσπάθεια που αλληλέγγυα προσπαθούμε να κάνουμε. Thank you very much. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής από την Γερουσία της Ρουμανίας. ο πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προφέρω καλά, ούτε καν να διαβάσω καλά. Μην ανησυχείτε, είναι, τα ρουμανικά ονόματα είναι δύσκολα, είναι γνωστό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το διπλό και το εξαπλό πακέτο σε στενή σχέση με τη συνθήκη περί δημοσιονομικής ε, εξυγίανσης γιατί αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντική για το άμεσο μέλλον. Και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη διοργάνωση αυτή της συζήτησης γιατί πρέπει να ομολογήσω πως στις χώρες μας δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ίσως θα μπορούσαμε έτσι να διευκρινίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της συνθήκης που δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές. Για παράδειγμα, τι σημαίνει που λέει medium round στο άρθρο 3 η... πώς λειτουργεί η διαδικασία στο άρθρο 7. Αλλά εγώ θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα. Ε, αυτή η συνθήκη είναι σημαντική διότι προωθεί δύο νέους ε, δείκτες κλειδιά που δεν έχουν οριστεί όμως πολύ καλά. Το πρώτο είναι το διορθωτικό έλλειμμα. Παρακολουθώ ε, τα στοιχεία από το Συμβούλιο και την Κομισιόν για το διευθυντικό έλλειμμα ε, της κάθε χώρας. Για τη χώρα μου, για παράδειγμα, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για το 2008-2009 γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ διαφορά ανάμεσα στην αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαίνει πως η μεθοδολογία που ακολουθείται δεν είναι σαφής. Αν μιλάμε για 0,5 έλλειμμα, θα πρέπει να ενοποιήσουμε τις ε, μεθοδολογίες έτσι ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεύτερη παρατήρηση. Ο πιο σημαντικός δείκτης είναι το δυνητικό ΑΕΠ, διότι όλα λειτουργούν γύρω από αυτή την έννοια κλειδί. Δυνητικό ΑΕΠ. Και κενό παραγωγής, χάσμα παραγωγής, output gap. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, εάν λάβουμε υπόψη το 2% δυνητικό ΑΕΠ, τότε ε, ε, θέτουμε σε κίνδυνο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας μας για το μέλλον. Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να ε, αυξηθούν οι προσδοκίες και να μειωθούν τα κενά ανάμεσα στην χώρα μου και τις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ένωσης. Και δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει αυτό με αυτές εδώ τις διατάξεις. Όταν συζητάμε λοιπόν για αυτό το Fiscal Compact, λάβατε υπόψη σενάρια, πιθανότητες αντικτύπου για κάθε χώρα, για το πώς δηλαδή αυτή η συνθήκη θα λειτουργήσει και ποιες θα είναι οι συνέπειες σε σχέση όχι μόνο με την ονομαστική σύγκληση, αλλά την πραγματική σύγκληση ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής θα είναι από τη Βουλή των Κοινοτήτων, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριος Κάσ. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Η δική μου ανησυχία για όλα αυτά στρέφεται γύρω από τον εξαναγκασμό επανέρχομαι σε κάποια σχόλια που έκανα πριν. Εγώ βρίσκω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για τις Εθνικές Βουλές. Και δεν περιορίζονται βέβαια μόνο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, οι ανησυχίε εννοώ, σχετικά με την επιβολή φόρου στις δαπάνες, που είναι προνόμιο του Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι πολίτες εκλέγουν ακριβώς γι' αυτό του εκπροσώπου τους στα κοινοβούλια, στις γενικές κοινοβουλευτικέ εκλογές. Εξετάζω τα έγγραφα εδώ, το έγγραφο μάλλον που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω αν κανεί άλλο το έχει διαβάσει, αλλά εδώ μιλούν για την European Financial Conference και λένε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκες πολιτικές διαπραγματεύσεις για να δοθεί το δημοσιονομικό καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τι λένε, κοιτάξτε παρακαλώ. Το παράδειγμα, ας πούμε, των υπουργών, των εθνικών υπουργών, από τους οποίους θα αναμένεται να μαρτυρούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποχρεώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταθέτουν δηλαδή, και βάζει και μια φράση ακόμη, οι εθνικοί υπουργοί μπορούν να θεωρούνται υπόλογοι μόνο στις εθνικές βουλές. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ εν πάση περιπτώσει. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι μέσω του μηχανισμού της έκδοσης νόμων με τρόπο φοβούμε ε, στην ουσία αντιδημοκρατικό δεν μίλησα ακόμη για ε, ειδικέ πλειοψηφίε, λαμβάνονται μέτρα για συντονισμό των φορολογικών πολιτικών που όπως είπα είναι αποκλειστικά, αποκλειστικά αρμοδιότητα των Εθνικών Βουλών. Άρα λοιπόν εδώ πρώτο ερώτημα που ανακύπτει. Το δεύτερο είναι ότι ο εξαναγκασμός που παρακολουθούμε σε σχέση με την περίπτωση της Ελλάδας όσα ελλείμματα και αν έχει σχετικά με το πώς τα καταφέρνει οι λόγοι, οι αιτίες και το ότι τις επέτρεψαν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 90 ενώ πολλοί πιστεύουν ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να έχει μπει η Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ο μιλητής. εγώ αγαπώ την Ελλάδα αλλά φοβούμαι ότι οι περιστάσεις υπό τις οποίες έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και ο ρόλος ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην αγορά αλλά και αποφάσεις που έλαβαν επιμέρους χώρες όταν συμφώνησαν, αποτελεί ένα πρόβλημα που τώρα βέβαια φαίνεται καθαρά. Ο εξαναγκασμός, επαναλαμβάνω, που οδήγησε στο πώς θα επιληθεί το οικονομικό χάος που έχει προκύψει από όλες αυτές τις συνθήκες, επίσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και που οδηγεί σε υπουργούς τεχνοκρατικών κυβερνήσεων που δεν έχουν πραγματικά εκλεγεί και που αυτοί χειρίζονται τώρα τα οικονομικά και πάλι εδώ νομίζω ότι δεν με έπεισε ο κ. Μπαρόσο λέγοντας ότι έχει εκλεγεί ο ίδιος με τον τρόπο που εκλέγεται τέλος πάντων. Εν τέλει θα πω το εξή. Οι οικονομικές μέθοδοι που εφαρμόζονται δεν είναι θέμα μεθοδολογίας, είναι θέμα του πώς λειτουργεί η διαδικασία στην πραγματικότητα. Ουδής εξετάζει τους λόγους και τι αιτίε που τα πράγματα πήγαν στραβά και φοβούμε ότι το πρόβλημα της αναπτύξεως δεν πρόκειται να λυθεί εάν δεν υπάρξει ελευθέρωση αυτή η deregulation και να δοθεί περισσότερο οξυγόνο, ζωή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θα προσθέσω απλά ότι το να ζητούμε όλο και περισσότερο να μαζεύουμε λεφτά είναι υποκατάστατο του τραπεζικού συστήματος που ναι μεν σωστά επικρίνεται αλλά με τους διάφορους φόρους για ε, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές κτλ. δεν θα έχουν καμιά επίπτωση θετική στην ανεργία των νέων που είναι τεραστία σε ορισμένες χώρες μέλη. Φοβούμε ότι θα δούμε περισσότερες διαδηλώσεις, περισσότερη αταξία, αύξηση στην δύναμη της άκρας δεξιάς, ενδεχομένως και της άκρας αριστεράς, δεν ξέρω, αλλά όταν θα συζητήσουμε και τη συνθήκη αύριο που υποτίθεται θα οδηγήσει σε συντονισμό και ανάπτυξη. Φοβούμε ότι θα οδηγήσει περισσότερο σε αποδυνάμωση των κυβερνήσεων, περισσότερη περισσότερες αντιθέσεις και πολύ φοβούμε ότι θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπίσουμε πρακτικά το πρόβλημα ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για έλλειψη δημοκρατία. και φοβούμε ότι δεν υπάρχει απολύτω καμιά ένδειξη από την συνάντηση μέχρι τώρα όπω παρακολουθώ αυτή τη διάσκεψη τώρα ότι κανεί εδώ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν τις πραγματικά υπάρχουσες συνθήκες. Έχω ακόμα μερικούς πριν δώσω την δυνατότητα να απαντήσετε. Από τη Λιθουανία λοιπόν, ο κύριος Γκλαβέκας της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου τους. Αν είναι παρόν. Okay. Καλά λοιπόν θα τον αφήσω στην άκρη, μήπως επανέλθει. Τσεχική Δημοκρατία, Γερουσία, ο κ. Σεύτσιτς, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στην σημερινή συνεδρίαση. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να συζητούμε και στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΣΑΚ, καθώς και σε διάφορες συνεδριάσεις και συναντήσεις μάλλον εθνικών βουλευτών με ευρωβουλευτές. Εγώ πάντως είμαι πολύ υπέρ της ιδέας αυτής της ΚΟΣΑΚ. Βρίσκομαι εδώ υπό διπλή ιδιότητα. Εκπροσωπώ το κυβερνών κόμμα, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερουσία, που δεν έχει όμως πλειοψηφία, και να πω λίγα λόγια για την τσεχική δημοκρατία. Όπως ξέρετε, η τσεχική δημοκρατία δεν υπέγραψε το λεγόμενο Fiscal Compact. Παρ' όλα αυτά, έχουμε νομοσχέδιο το οποίο θα μας οδηγήσει στην ίδια κατεύθυνση της δημοσιονομικής πειθαρχία. Είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια τώρα στην τσεχική δημοκρατία και που άρχισε πριν από την ελληνική κρίση. Ήδη το 2000 είχαμε αρχίσει να έχουμε σημαντικά προβλήματα εμείς στον δικό μας τραπεζικό τομέα Ορισμένες από τις τράπεζές μας είχαν συσσωρεύσει πολύ υψηλά χρέη και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά ήδη πολύ νωρί. Ίσως ορισμένοι από εσά μπορείτε να αντλήσετε κάποια διδάγματα από τα όσα πράξαμε τότε. Ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά οδυνηρή. Δεν ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ΕΚΟΦΗΝ να μας βοηθήσουν. Καταφέραμε μόνοι μας να ξεπεράσουμε την κρίση εκείνη και τα καταφέραμε μάλιστα να βοηθήσουμε και άλλες χώρες μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχω ζήσει χρόνια πολλά σε σχεδιαζόμενη οικονομία, κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία και όπως ο προλαλής σας κύριος Κάσ, έχω και εγώ ορισμένε επιφυλάξεις. Δεν θέλω το ευρωπαϊκό εξάμεινο να υπαγορεύσει στις χώρες μέλη πώς θα σχεδιάσουν τις οικονομίες τους, διότι αυτό θα μας στερήσει ένα από τα σημαντικά πλονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του ανταγωνισμού. Ποιος προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να λύσει την κρίση. Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ή όποιοι το χρειάζονται αυτό. Πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Και αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική της Ευρώπης 2020 πρέπει να είναι περισσότερες δουλειές ανάπτυξη βασισμένη στην επιστημονική πρόοδο. Αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Πρέπει να απαλείψουμε τους φραγμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ενιαία αγορά και που είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα, η αγορά δηλαδή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χαρεί πολύ με μερικά ευρώ που θα μαζέψει ακόμα από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει εκεί μεγάλο μέλλον. Ούτε μου αρέσει πολύ η ιδέα της επιβολής φόρου στους πλουσίους. Δεν έχω πρόβλημα να συζητούμε τα θέματα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φορολογούμε τους επιτυχημένους. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις. Η Ιρλανδική Βουλή, Τόμας Μπέρν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες σκέψεις για την κατάσταση στην Ιρλανδία και την εμπειρία που έχουμε από τότε που προσχωρήσαμε στο ευρώ. Αξίζει να πούμε ότι θα ήμασταν εν πλήρη συμμορφώσει με το Fiscal Compact ε, από την αρχή του ευρώ μέχρι και το 2008, όπου ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και φάνηκε ότι διαχειριζόμασταν λάθος την οικονομία μας και αυτό ήταν προφανές τελικά. Είναι σημαντικό δηλαδή να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη αυτό που είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι δηλαδή πρέπει να επανέλθουμε στην οικονομική ανάπτυξη, να δώσουμε προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας και κυρίως της ανεργίας των νέων. Είναι βασικό θέμα συζήτηση στην Ιρλανδία όπως και στη Ρουμανία, ε, λόγω ε, της ισχύς που έχει το δημοψήφισμα ως προς την επικήριση του Fiscal Compact. Η ευρωπαϊκή οικογένεια φαίνεται να είναι μια οικογένεια που ενδιαφέρεται κυρίως για την επιβολή της πειθαρχίας και της δημοσιονομικής λιτότητας και αυστηρότητας, χωρίς να δίνει σημασία στο θέμα της ανάπτυξης και της ανεργίας. Έχουμε φορολογικούς ελέγχους, αλλά δεν έχουμε φορολογική ένωση και έτσι δεν έχουμε τα ωφέλη που θα είχαμε από τη φορολογική ένωση, τα εμβάσματα, τις μεταφορές, πράγματα που ως Ιρλανδία θα ε, είχαμε αξιοποιήσει. Από εκεί και πέρα, η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αυστηρότητα των ελέγχων από τη μία χωρίς φορολογική ένωση από την άλλη είναι ακριβώς η αιτία που έχει οξύνει τα προβλήματά μας ως χώρα και ως εθνική οικονομία. Πολλές από τις διατάξεις και πολλές από τις διαδικασίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολλά σημαντικά πράγματα. Στη διάδα των μέτρων η υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού είναι μεν σημαντική, ωστόσο συνεπάγεται σημαντική αλλαγή στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούσε σε αυτή τη συνθήκη, γιατί εμείς έχουμε διαφορετική διαδικασία. Ήμασταν ανέκαθεν εξαιρετικά δημοκρατικοί στη διαδικασία αυτή όλος ο πολιτικός κύκλος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα εστιάσει την προσοχή του στο ε, προϋπολογισμό και θα γίνονται διάφορες ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και αυτή η δυνατότητα μειώθηκε με τα καινούργια μέτρα. Οι προτάσεις για την αύξηση του ΦΠΑ πέρσι ακούστηκαν για πρώτη φορά στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν να φτάσουν στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, παρόλο που ο ΦΠΑ ε, αφορούσε τη δική μας χώρα. Η ψήφιση του προπολογισμού είναι ε, μια ε, εν το δημοκρατική διαδικασία και δεν μπορούμε να τη χάσουμε γιατί έτσι οι Ιρλανδοί θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ ο κύριος Βαλεντίν Νικολόφ από την ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο έδωσε εντολή στην κυβέρνησή μας να διαπραγματευτεί και να υπογράψει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Υπό έναν όρο, να μην οδηγήσει αυτό σε φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην υπάρξει ε, φορολογική εναρμόνιση και εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών. Στην Βουλγαρία ήδη από το 2010 ε, τροποποιήθηκε η νομοθεσία περί του προϋπολογισμού και τώρα έχουμε την οροφή του 2%. Το έλλειμμα ανέρχεται στο 33,5% του ΑΕΠ και μάλιστα ακόμα και πριν να συζητηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας στη Βουλγαρία, η κοινωνία μας ήδη συζητούσε ορισμένα μέτρα ήδη τα είχε αποδεχθεί και ε, καταλήξαμε ε, σε μια κοινή γραμμή στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας και δεν θα είμαστε σε θέση υπ' αυτή την έννοια να επιτύχουμε τους στόχους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Ακόμα και πριν από την κρίση, ακόμα και πριν από το 2008, εμείς ως χώρα είχαμε μια σωστή φορολογική πολιτική και έχουμε μειώσει το έλλειμμα για το 2011. Για το 2011 το έλλειμμα θα ανέλθει στο 1,3%. Το χρέος φτάνει στο 19% Όλα αυτά τα οποία προβλέπονται θα αυξήσουν το βάρος που επομίζονται οι Βούλγαροι πολίτες. Ένας από τους βασικούς μας εταίρους, η Ελλάδα, διανύει περίοδο βαθιάς ύφεση. Επομένως, η Βουλγαρία θα πρέπει να προσπαθήσει να αναδιαρθρώσει την οικονομία της και θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα για τη μείωση του εισεζυγίου ε, τρέχουσών πληρωμών. Αυτή τη στιγμή σημειώνουμε πλεόνασμα της τάξης του 1,5%. Το ερώτημά μου είναι το εξής πέρα από τους μηχανισμούς για τις απειθάρχητες χώρες, μήπως θα έπρεπε να βρούμε και τρόπους να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τις χώρες που έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχία. Γνωρίζετε πολύ καλά πιστεύω ότι ό,τι φορολογικά μέτρα, όποια φορολογικά μέτρα και αν υιοθετήσει κανείς, δεν έχει ουσιαστικά επαρκή μηχανισμό ή τουλάχιστον στη Βουλγαρία δεν υπάρχει επαρκής μηχανισμός για να ενθαρρύνει ουσιαστικά την ανάπτυξη. Θεωρείται η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή ως μία από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο ανάπτυξης. Δεν φτάνει όμως αυτό. Μας χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη. Επομένως μέτρα ενθάρρυνσης των χωρών που έχουν δημοσιονομική πειθαρχία θα ήταν κάτι το εξαιρετικά θετικό χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια για το τι θα συμβεί ε, στην περίπτωση κατά την οποία τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα δεχθούν τα μέτρα που, προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτός στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Θα ήθελαμε να απαντηθούν αυτά τα ερώτηματα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ η Σιλβή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάποιος άλλος ενδεχομένως μπορεί να απαντήσει από την αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι κρίμα που έφυγε ο κύριος Κάς, γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε να αποφύγουμε, να μην συζητάει ο ένας με τον άλλον. Εγώ ήμουν η του κειμένου με τη στήριξη των συναδέλφων, του κειμένου που είχε να κάνει με τον οικονομικό διάλογο και ο σκοπός του οικονομικού διαλόγου αυτού που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ απλός. Οι οικονομολόγοι θα έλεγαν ότι σκοπός του οικονομικού διαλόγου είναι να λάβει υπόψη του τις εξωτερικές διαστάσεις και επιπλοκές των εθνικών πολιτικών. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει φόρουμ, μέρος αν θέλετε, όπου μπορούμε να συζητήσουμε, να συζητήσουμε απλά και μόνο, χωρίς έλεγχο, χωρίς λογοδεσία για οικονομικά θέματα. Μόνο οι Υπουργοί Οικονομικών το μόνο που να κάνουν να έρθουν εδώ και να εξηγήσουν τι κάνουν στις χώρες τους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι φοβάστε, ε, ζητώ από σας να ρωτήσετε τον κύριο Κάσου, τι φοβάται εν πάση περιπτώσει, γιατί πιστεύει ότι η δημοκρατία, η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει πάντοτε να είναι αυστηρά περιχαρακωμένο σε εθνικό πλαίσιο. Σήμερα σήμερα που ο κόσμος μας είναι πολύ περισσότερο αλληλεξαρτημένος από ό,τι παλιά. Εάν λάβουμε εμείς εσφαλμένες αποφάσεις μπορεί να καταρρεύσει το σύντη του Λονδίνου. Εάν η Βροζώνη κάνει κάποιο λάθος, ίσως εσείς θα πρέπει να ε, υποστείτε τις συνέπειες. Αυτό είναι ο μόνος σκοπός του οικονομικού διαλόγου, για να επιστρέψετε δηλαδή στις επατρίδες σας και να εξηγήσετε ότι ε, θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε πώς ακριβώς είναι ο κόσμος μας. Ένας κόσμος με όλο και περισσότερες αλληλεξαρτήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βάσει συνθήκων κυρωμένων και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ε, συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ ε, που μου δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Δυστυχώς εν τη επουσία του βουλευτή που ασκεί κριτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Μιριέλ Κέρκενς από το Βέλγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η χαίρομαι ιδιαίτερος διότι έχουμε την ευκαιρία να διεξάγουμε αυτή την κοινή συζήτηση όλοι μας εδώ σε αυτή την αίθουσα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που είμαι μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βέλγιο. Εν πάση περιπτώσει στο Βέλγιο ξέρετε ότι είμαστε όλοι υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μιας όσο ε, των περισσότερο ενοποιημένη πολιτική, η οποία βέβαια πάντοτε θα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Υπ' αυτή την έννοια δεν θα διαφοροποιηθώ από τους συναδέλφους. Σε σχέση με το έργο τώρα που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την δουλειά των εισηγητών, ως μέτρο προφύλαξης σε αυτά τα δύο σχέδια κανονισμών θα ήταν καλό να συμπεριληφθεί μια πρόβλεψη βάσει της οποίας θα γίνεται σεβαστός ο τρόπος διαβούλευσης από πλευράς κράτους με τους κοινωνικούς του εταίρους, π.χ. σε θέματα μισθολογικά. Δηλαδή, να, ε, μπορεί το κράτος να έχει την ευχαίρεια π.χ. να οργανώσει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια στη χώρα αυτή, χωρίς να ε, τίθενται ένα αμφιβόλο ή να διακινδυνεύουν ε, λόγω δικτών, λόγω μηχανισμών εποπτείας που θα αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως είναι αναγκαίο να εξετάσουμε την χρονική συγκυρία και να ε, επιτρέψουμε ε, την ευκαιρία για διαβούλευση, για συνδιαλλαγή. Και από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τους προϋπολογισμούς των ε, κρατών, καλό πάντοτε θα ήταν να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων ε, και μάλιστα σε ομοσπονδιακά κράτη αυτό είναι πολύ πιο απαραίτητο. Ε, θα πρέπει η χρονική συγκυρία λοιπόν να ε, εξεταστεί με σοβαρότητα. Και βεβαίως οι κοινωνικές διαστάσεις, τα θέματα τα περιβαλλοντικά, η καταπολέμηση της ανεργίας η ενίσχυση της απασχόλησης δεν θα πρέπει να παραμελούνται ε, προς όφελος της ε, δημοσιονομικής πειθαρχία. Συν της άλλης, θα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ε, και βάσει της οποίας εκδίδει γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης για την κατάσταση κάθε χώρας και γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στο, στις διορθώσεις που θα πρέπει να επιβάλλει το συγκεκριμένο κράτος. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι το εξής. Αν ένα κράτος έχει ακολουθήσει τις συστάσεις και συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, να μην θεωρείται υπεύθυνο γι' αυτά από τη στιγμή που ακολούθησε κατά γράμμα τις συστάσεις. Και θα ήθελα και περισσότερες εξηγήσει ως προς αυτό που είπατε ε, όταν ένα κράτος βρίσκεται στο όριο κήρυξης τάσης πληρωμών να μπορεί να απολαμβάνει μιας νομικής αφήνειας, αν θέλετε, βεβαιότητας όπως μια επιχείρηση. Μπορείτε αυτό να το διευκρινίσετε περαιτέρω. Και ως προς το σχέδιο κανονισμού που έχει να κάνει με την εποπτεία των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είναι σημαντικό να απαιτήσουμε να οριστούν καλύτερα αυτές οι σοβαρές δυσκολίες οι οποίες ε, μπορεί να εντοπιστούν. Περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν οι δυσκολίες ως σοβαρές. Τι θα συμπεριληφθεί σε αυτόν τον ορισμό. Συμφωνώ βεβαίως με την ανάγκη ε, συγκρότησης ενός ταμείου που θα βοηθήσει τα διορθωτικά ταμεία για να υπάρξουν επενδύσεις στις υποδομές. Και είναι βεβαίως καλό το γεγονός να μπορεί το Συμβούλιο Υπουργών να παρεμβαίνει πέρα από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερωτώ όμως, ποιο είναι το περιθώριο ελιγμών που υπάρχει στις συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου ως προς το σχέδιο κανονισμού. Αυτά τα δύο σχέδια κανονισμών. Άπαξ και ενσωματώσουμε τις διατάξεις στον κανονισμό αυτό, τότε τι νόημα έχει να υπάρχει αυτή η συνθήκη ε, του Fiscal Compact. Ε, αν ενσωματωθούν στους κανονισμούς οι διατάξεις, ε, ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτής της συνθήκης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Στη συνέχεια, ο κ. Τζιανκάρλο Τζοτζέτη, Πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, θεμάτων προϋπολογισμού της Ιταλικής Βουλής. Παρακαλώ. Grazie. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θεωρώ και υπό το φως της Ιταλικής εμπειρίας ότι σίγουρα είναι χρήσιμο μέσο, αλλά ίσως δεν καταφέρνει να λάβει πλήρως υπόψη την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι επίγουσες καταστάσεις κινδυνεύουν να ταράξουν εντελώς τις προβλέψεις που γίνονται ετησίως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ιταλίας, για παράδειγμα, το πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλησης που κατά κάποιο τρόπο είχε οριστεί την περασμένη άνοιξη τελείως ανατράπηκε και μάλιστα ξεκίνησε μια, ένα άλλο είδος πολιτικών, όχι μόνο λόγω της απειλής επιβολής κυρώσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την ε, κρίση των αγορών. Πιστεύω πως οι χρηματοπιστωτικές αγορές δίνουν μια εξολόγηση όσον αφορά τα spread σχέση με τους γερμανικούς τίτλους, ας πούμε, στην δική μας ε, περίπτωση, που οδήγησαν την κυβέρνησή μας να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή μια αξιολόγηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πολύ πιο πριν και πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη πίεση έρχεται η αξιολόγηση από τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Ίσως ε, ε, αυτό το θέμα του οργανισμού αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να εξεταστεί. Η Ιταλία έχει ακολουθήσει μια πορεία δημοσιονομικής πειθαρχία τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να κάνει την ίδια προσπάθεια. με πρόβλημα πολύ ψηλού ελλείμματος πολύ ψηλού χρέου και του επόμενου μήνε θα εγκρίνουμε την συνταγματική μεταρρύθμιση για την ε, ένταξη του ισολογισμού και, της, ε, και της, ε, των σχεδίων προπολογισμών, της εποπτείας μάλλον του προϋπολογισμού. Θα γραφεί όλο αυτό μέσα στο Σύνταγμα. Εγώ θα ήθελα να έχω κάποιες διευκρινήσει, αν μπορείτε να μου τις δώσετε. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τον ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης σε σχέση με την παρακολούθηση και την εποπτεία αυτού του σχεδίου προπολογισμού. Θα είναι ένα ανεξάρτητο οργανισμός που θα λειτουργεί παράλληλα με το Κοινοβούλιο και... Βεβαίως μιλήσαμε για δημοσιονομική λιτότητα αλλά είναι κάτι άλλο η συνταγή της ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω πως οι ιδιαιτερότητες των οικονομιών μας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια ενιαία απάντηση, μια ενιαία συνταγή. Δεν πιστεύω, ας πούμε, όσον αφορά τις πιστώσεις, τα έσοδα, που, μάλλον οι συνταγές που υποδεικνύονται, θα έχουν την ίδια απόδοση σε διαφορετικά συστήματα. Γιατί το αγγλοσαξονικό, για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετικό από το ιταλικό που βασίζεται σε μικρές ε, τράπεζες ε, εταιρικού τύπου και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ από την Εστονία ο κ. Στάβη Ρόιφες που είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο στην, τελευταία, στην προηγούμενη συζήτηση ακούσαμε πως η Φιλανδία ήταν μια από τις χώρες που είχε ισορροπημένο, ισολογισμένο μάλλον προϋπολογισμό ακόμα και πριν από την κρίση και κατά τη διάρκεια αυτής. Αυτό ισχύει όμως και για την Εστονία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία. Ε, εντάξει, η Σουηδία... Βέβαια είναι στην, έχει ακόμα τη Σουηδική κορώνα, αλλά είναι υποδειγματική όσον αφορά την ε, διαχείριση των οικονομικών της. Τέσσερις από τους 27 όμως δεν αρκούν Το να βάλει κανείς τάξη στα οικονομικά του είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη οικονομία και οι τέσσερις αυτές χώρες είναι επιτυχημένες οικονομικά. Όλοι πρέπει να μπορούν να φροντίσουν τα χρήματά τους και κυρίως τα χρήματα των φορολογουμένων. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια χώρα με 30% υψηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλήν από ότι η Εστονία, όπου τη μισθή είναι διπλάσια από του δικούς μας. Δεν νομίζω όμως πως κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο και εδώ για βιωσιμότητα πρόκειται. Την περασμένη Πέμπτη αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο να στηρίξουμε αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι διαρθωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις Έχουμε μια ευκαιρία τώρα, εν μέσω της κρίσης, να κάνουμε τις διαφορετικές αλλαγές που χρειάζονται και οι ψηφοφόροι καταλαβαίνουν καλύτερα το τι κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, είναι όμως διαφορετικές. Δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση ενιαία. Αν δούμε όμως τα στοιχεία, υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην ορθή ε, δημοσιονομική διαχείριση, την απλή ε, διάρθρωση της φορολογίας και την οικονομική επιτυχία. Γνωρίζω χώρες που έχουν επιτύχει έσοδα, όχι αυξάνοντας τους φόρους, αλλά μειώνοντας τις εξαιρέσεις. Νομίζω πως αξίζει να ανταλλάξουμε τέτοιου είδους εμπειρίες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και περνάμε στην Φιλανδία και τον Κίμο Σάση που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η κρίση χρέους στην Ευρώπη είναι πολύ λυπηρή ιστορία. Ο λόγο ε, στον οποίο οφείλεται η κρίση είναι ότι έχουμε τέσσερι κενσερνού προφήτες που ήρθαν και είπαν ότι τώρα στην οικονομική κρίση πρέπει να δαπανίσουμε και να δαπανίσουμε. Οι πολιτικοί το πίστευσαν και γι' αυτό βρεθήκαμε στην κρίση. πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε δύο προβλήματα στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι ότι δεν επικρατούν τα σωστά επιτόκια για τις σωστές χώρες. Το 2000 έπρεπε το επιτόκιο στην Ελλάδα να ήταν στο 8%. Συγγνώμη, το 2008 και να χαμηλώνουν τα επιτόκια ε, δεν είναι σωστή λύση. Μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή, αλλά ε, επιφέρει κινδύνους για το μέλλον. Και αν δούμε τι κάνει η Κομισιόν, όταν προσπαθεί να εισάγει τα ευρωομόλογα με χαμηλά επιτόκια για όλες τις χώρες, ούτε αυτό είναι ρεαλιστικό. Και μπορεί να αποτελέσει πηγή για περισσότερους κινδύνους και να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Κομισιόν δεν καταλαβαίνει όμως πού είναι τα προβλήματα. Το δεύτερο ε, ε, ακούστηκε μια καλή πρόταση από την Κομισιόν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό αξιολόγησης ε, των χρηπιστοληπτικής ικανότητας σε ευρωπαϊκό. Και θα έλεγαν, ας πούμε, θα, τους, θα την έφτιαχναν τον οργανισμό αυτό ή η Κομισιόν και θα έλεγε ναι, να δώσουμε επιστώσει στην Ελλάδα εκεί όπου χρειάζεται, όμως θα πρέπει κανείς να δει την πραγματικότητα και όχι να αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του. Δεύτερο είναι η διαφορά μεταξύ του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωμών στις διάφορες χώρες. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Και έπειτα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει χρήματα ή μεταφέρει χρήματα από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε άλλες και δεν υπάρχουν μηνύματα προειδοποιητικά. Πρέπει να βρούμε κάποια τέτοια σημάδια. Όταν δηλαδή το ισοζύγιο πληρωμών κάποιες χώρες δεν είναι ε, ε, σωστό. Πρέπει να πάμε δηλαδή στον πυρήνα της κρίσης και όχι να τρέχουμε διαρκώς και να προσπαθούμε απελπισμένα να λύσουμε την κρίση με οποιοδήποτε τρόπο. Ωστόσο, οι προτάσεις που αφορούν τον δημοσιονομικό έλεγχο και την υποπτία των χωρών που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες είναι σωστά βήματα. Όμως, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει και εκεί που δεν λειτουργήσε θα έπρεπε να έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ γραφειοκρατικό, αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά. Και ο στόχο είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και να σας πω ότι στη Φιλανδία είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα, ότι δηλαδή έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο τετραετές και Μετά από τέσσερα χρόνια θέλουμε να δούμε, ε, ελέγχουμε κατά πόσο η ισορροπία υπάρχει. Ε, δηλαδή, ο πιο μακρόχρονος προγραμματισμός βοηθά για να μπορεί κανείς να χειρίζεται σωστά την οικονομία του. Και όταν βλέπουμε την Κομισιόν, όλα είναι πολύ γραφειοκρατικά, έχουμε όμως περιορισμένους πόρους. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η Κομισιόν να θέσει σαφείς προτεραιότητες στο έργο της. Για παράδειγμα, δούμε διάφορε χώρε που δεν έχουν έλλειμμα. Εντάξει. Βλέπει κανεί μια χώρα και συζητάνε όλες οι χώρες, αλλά μετά η Κομισιόν δεν ε, αναμειγνύεται πολύ εκεί, γιατί δεν χρειάζεται. Οι χώρε όμω που έχουν προβλήματα θα πρέπει να τι εξετάζει πιο προσεκτικά η Κομισιόν. Ωστόσο, υπάρχει ε, σύγκρουση ανάμεσα στον εθνικό προπολογισμό και τις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθούν οι σωστοί τρόποι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι εμπίπτει στι εθνικέ αρμοδιότητε και τι στι ευρωπαϊκέ. Έπειτα αναφέρθηκε το 0,5%. Πώς μπορεί κανείς να το υπολογίσει αυτό. Ελπίζω να μην είναι μια διαρκής ε, ιστορία για το πόσο καλά είναι τα κριτήρια ή όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ξέρει κανείς περίπου που πηγαίνει και όλοι να κατανοούν ότι πρέπει να γίνουν διορθώσει όταν κανεί δεν πληρεί τα κριτήρια. Και οι χώρε οι οποίε δεν έχουν πρόβλημα μπορούν να φτάνουν στο έλλειμμα του 1%. Αυτό λέει ότι αν κανείς φροντίζει τα του οίκου του δεν χρειάζεται μεγάλη ανάγκη για υποπτία. Ωστόσο είναι πάντοτε πολύ καλό να συζητάμε και να παίρνουμε τις συμβουλές της Κομισιόν γιατί υπάρχει πολύ οικονομική γνώση και πυρογνωμοσύνη εκεί παρά τα όσα είπα στην αρχή. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής από την Σλοβενία είναι ο κύριος Σετσέβιτς που είναι ε, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική είναι πολύ χρήσιμο να συζητούμε με εκπροσώπους άλλων χωρών. Είναι αλήθεια. Για τη Σλοβενία ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία η Σλοβενία για πολλά χρόνια διεξήγαγε επιτυχημένες οικονομικές πολιτικές με χαμηλά χρέη, χαμηλό δημόσιο χρέος. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται η κρίση να έπληξε τη Σλοβενία σκληρότερα από άλλες χώρες μέλη, κυρίως διότι διπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος μας, αν και εξακολουθεί να περιμένει μέσα στα πλαίσια των κριτηρίων. Και το χρέος μας αυξήθηκε και το έλλειμμα. Τώρα, η νέα κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα πρόγραμμα για την εξυγένση των δημοσίων οικονομικών. Το 2012 οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα οδηγήσουν σε ένα μέγιστο, ένα maximum, δηλαδή 3% δημοσιονομικού ελλείμματος, που θα σημάνει βέβαια σημαντική λιτότητα για να επιτευχθεί, αλλά θα λάβουμε μέτρα και αντιστάθμισης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, δηλαδή τα υψηλά μισθολόγια θα μειωθούν, το ίδιο θα ληφθεί μέρημνα για το τραπεζικό μας σύστημα να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δώσουν περισσότερα δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι που είναι σημαντικό και νομίζω πρέπει να το πω εδώ και είναι σημαντικό ίσως και για άλλες χώρες μέλη είναι ο χρυσός αυτός δημοσιονομικός κανόνας. Ο χρυσός αυτός κανόνας θα ενταχθεί στο Σύνταγμά μας, αλλά αυτό προκαλεί ορισμένα ερωτηματικά. Δηλαδή πώς θα θεσπιστεί, πώ θα μπει στο συνταγματικό κείμενο ο χρυσό αυτό κανόνα. Κάτι όμως που έχει κάνει και η Ομοσπονδιακή Γερμανία και η Ελβετία και οι Ενωμένε Πολιτείε σε ένα βαθμό εφαρμόζουν το χρυσό αυτό κανόνα. Είναι όμως δύσκολο να γίνει και κυρίως σε ό,τι αφορά το ύψος του χρέους οι ορισμοί που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή Γερμανία και η Ελβετία είναι παρόμοιοι μεταξύ τους, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστούμε ένα ενιαίο ορισμό για όλους. Το επόμενο θέμα που ανέκυψε και όπου θα χρειαστούμε και από εσά κάποιες συμβουλές είναι το εξή. Δεν είναι μονάχα η Νομισματική Ένωση που ακούγεται τελευταία, αλλά και η Δημοσιονομική, η Φορολογική, αν θέλετε, Ένωση ακούγεται επίση. Πολύ, είναι πολύ επιφυλακτική. Πάλι εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει Δημοσιονομική Ένωση. Έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν. Ένας τρόπος είναι εναρμόνιση του φόρου επί των εταιριών και του ΦΠΑ. Αυτά είναι θέματα που αντιμετωπίζει βέβαια η Σλοβενία όπως και άλλες χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Είχε προβλεφθεί να προχωρήσω εγώ σε μια σύντομη σύνοψη, αλλά υπάρχουν ερωτήσεις ειδικώ για τους εισηγητέ. Θα προτείνω λοιπόν να λάβουν το λόγο σύντομα οι εισηγητέ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, κυρίως αυτές που σχετίζονται με τις εκθέσεις τους και εγώ θα προσπαθήσω μετά να απαντήσω σε κάπως πιο γενικές ερωτήσεις. Ελίσσα, είχατε εσείς κάποιες πρώτες ερωτήσεις από Γάλλους συναδέλφους. Ναι, για να εξοικονομήσουμε χρόνο θα μιλήσω αγγλικά. Δύο ή τρία, τρία θέματα που αποτέλεσαν συγκεκριμένες ερωτήσεις προς εμένα ή σε σχέση πάντως με την έκθεσή μου. για το πρόβλημα της πραγματικής σύγκλησης και πώς να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί το διαθροτικό έλλειμμα. Βρίσκω ότι αυτό είναι σημαντικό, πραγματικό θέμα και, και θέμα μεθοδολογίας ειδικότερα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά για να υπάρξει μια κοινή συμφωνία, μια συνεννόηση από αυτού. Επίσης οι μακροοικονομικές ανισότητε, η διάσταση των μακροοικονομικών ανισοτήτων που είναι νέα διάσταση και προέρχεται από το λεγόμενο six pack, τη δέσμη των 6 μέτρων, να μας βοηθήσει δηλαδή να αντιληφθούμε πώς η ίδια η λειτουργία της ενιαία αγοράς προκαλεί τι ανισότητες αυτές μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο, για παράδειγμα, η Σουηδία, οι κάτω χώρε, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο εξακολουθούν και έχουν επιμόνως υψηλά πλεονάσματα, ενώ 20 χώρες έχουν μόνιμα ελλείμματα και ορισμένε και πάρα πολύ υψηλά. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε ποιε είναι οι αιτίε αυτών των ανισοτήτων μέσα από την ενιαία αγορά. Επίσης, τα προβλήματα της φορολογίας δεν μπορούν να μείνουν απ' έξω, καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν ορισμένες πολιτικές στους γείτονες, σε γειτονικές χώρες δηλαδή. Για τους λόγους αυτούς προσπαθούμε στο χρονοδιάγραμμά μας και έχουμε εδώ στην πρώτη ερώτηση ιδίω. η επιθεώρηση, η ετήσια επιθεώρηση ετήσιας ανάπτυξης να είναι πρώτη πριν από την δημοσίευση των ε, policy orientations από πλευράς Κομισιόν και Συμβουλίου μέσα στο ίδιο το εξάμεινο και αργότερα οι χώρες μέλη να έχουν επαρκή χρόνο και εμείς προτείνουμε να αλλάξουμε την 15η Οκτωβρίου ημέρα της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού στην 30 Σεπτεμβρίου, ώστε μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 30 Οκτωβρίου να υπάρχει περίοδος διαλόγου και επίσης ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει το σχεδιασμό, να, που, να εξτάσουμε το σχεδιασμό που υποβάλλουν διάφορες χώρες και στις 30 Νοεμβρίου να υποβάλει τη γνωμοδότησή της για το δημοσιονομικό σχεδιασμό η ε, Κομισιόν. Να μην περιορίζεται δηλαδή ο χρόνος ε, εξέτασης από την Κομισιόν περιορίζοντας έτσι την λειτουργία της δημοκρατίας και μέσα σε κάθε χώρα μέλος. Μπορώ να συζητήσω και με λεπτομέρειες τις προτάσεις αυτές, εφόσον το επιθυμείτε. Και το τελευταίο μου σχόλιο για τα ομόλογα σταθερότητας και το Ταμείο Διάσωσης. Αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει εκδώσει σχετικά ψηφίσματα και για την ε, Δημοσιονομική Συμφωνία, το Fiscal Compact, όπου το Κοινοβούλιο όμως δεν ήταν συνομοθέτης, ήταν μόνο παρατηρητής. Πάντως έχει εγκριθεί από πλειοψηφία το κείμενο αυτό από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες και στο κείμενο αυτό, στο ψήφισμα αυτό δηλαδή, το Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ένα συντονισμό με κατευθυντήρες γραμμές και όρους και ζητάει επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της νέας συνθήκης με τα ομόλογα σταθερότητας μέσα στα πλαίσια της πράσινης πίπλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το Ταμείο Διάσωσης. Αυτά δεν είναι ασύμβατα με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σταθεροποιητικού Μηχανισμού που επίσης στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι με λίγα λόγια νομίζω μέσα στα χρονικά περιθώρια που διαθέτω, ε, αυτές, μπορούν, αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορώ να δώσω στις ερωτήσεις που αφηθήθηκαν σε μένα ως εισηγήτρια, αλλά βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσω και διμερώς αν θέλετε μαζί σας ε, με περισσότερο χρόνο να συζητήσω με όλους τους βουλευτές που επιθυμούν να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις προτάσεις. Μια τελευταία λέξη για την κυρία Γκέρκενς. Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν για θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και βιωσιμότητα και για τις μακροοικονομικές. Ε, μάλλον μπαίνουν, στην έκθεση για τις ε, μακροοικονομικές ανισότητες και εκεί προσπαθώ να εξηγήσω πώς τα βλέπουμε για την ε, ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θεωρητικά βέβαια έχει λήξει ο χρόνος μας. Πολύ σύντομα λοιπόν παρακαλώ Ζαν ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους πράγματι, όλοι ε, έδειξαν ότι σέβονται ε, τις απόψεις των άλλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει στόχο να προσποριστεί τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέλουμε να ασκούμε δημοκρατικό έλεγχο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν θέλουμε καθόλου να ανακατευθούμε στις εθνικές υποθέσεις. Να απαντήσω στην ερώτηση της Βελγίδας συναδέλφου. Καταρχάς να πω ότι δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σας Το θέμα είναι η σύνδεση μεταξύ των συστάσεων και της δημοκρατικής ε, λειτουργίας του κράτους. Εδώ μπορούμε να προβληματιστούμε, να βρούμε λύσεις. Πώς ε, θα προλάβουμε και δεν θα δημιουργηθεί η αρνητική κατάσταση που περιγράφεται. Από εκεί και πέρα η διαδικασία της ασφαλιστικής δικλίδας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλούμε για το άρθρο 11. Δηλαδή, δεσμεύονται και παγώνουν οι αξιολογήσεις οι οποίες επηρεάζουν ε, τα επιτόκια, ε, παγώνουν τα επιτόκια σε συγκεκριμένο επίπεδο. Θα πρέπει επίσης οι πιστωτές να δηλώσουν την ιδιότητά τους αυτή μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό ε, διάστημα. Άλλωστε, ως προς την Ελλάδα, η, η κατανομή, η πολύ ευρία κατανομή του ελληνικού χρέους και η άγνοια για το ποιος το κρατά τελικά, ποιος το κρατούσε όλο αυτό τον καιρό, ήταν κάτι που δυσκόλευσε πολύ τις διαπραγματεύσεις. Όλες αυτές είναι οι προτάσεις που έχουμε, δηλαδή να ισχύσουν αυτά και για το κράτος όπως ισχύουν και για τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό επίσης ε, ε, θέλησα να συμπεριλάβω στο κείμενο την παρέμβαση του Συμβουλίου εκτός από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ορισμός των σοβαρών δυσκολιών και το περιθώριο ελιγμών που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να μην είναι πολύ περιορισμένο. Από τότε που ξέχασε η κρίση, είναι εξαιρετικά δύσκολε οι διαπραγματεύσει μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, διότι στο Συμβούλιο σπάνια υπάρχει μια πολύ ισχυρή ε, κοινή θέση και προσπαθεί η Προεδρία του Συμβουλίου να συμφιλειώσει του μεν και του δε, ενώ συνήθω το Κοινοβούλιο ε, μιλάει με μία φωνή ως προς τα θέματα αυτά. Ξέρετε, είμαι μεγάλος, ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κανόνας, ο χρυσός κανόνας, η διάταξη αυτή είναι μια διάταξη που θα μείνει στη συνθήκη, επομένως η συνθήκη έχει λόγο ύπαρξης κατά την άποψή μου. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο κανονισμών και ε, για τα περαιτέρω υπαρξιακά ερωτήματα μεταξύ ως προς τη συνθήκη θα ασχοληθούν οι έγκριτοι νομικοί. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στην, στον κύριο Κρέινερ, ο οποίος θέλει να απαντήσει για κάποια φορολογικά ζητήματα. Ναι, και εγώ θέλω να σχολιάσω ή να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Μεσοπρόθεσμος προπολογισμό και πρόγραμμα σταθερότητας. Ποιο είναι ε, μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ποια, ποια είναι διαφορά. Νομίζω ότι ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει ένα πρόγραμμα σταθερότητας το οποίο εφαρμόζεται όταν μια χώρα χρειάζεται επιπρόσθετα μέτρα. Ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός υφίσταται ούτως ή άλλως. Ε, εμείς στην Αυστρία τον εγκρίνουμε κάθε χρόνο. Κάθε άνοιξη ε, κάνουμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση, μια ενδιάμεση επισκόπηση της, του πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός. Και αυτή τη στιγμή συζητούμε περί ενός προγράμματος σταθερότητας. Και έτσι ε, η ενδιάμεση αναθεώρηση λαμβάνει υπόψη της θέματα του συμφώνου σταθερότητας. Τώρα έχουμε ε, μείωση της ανάπτυξης κατά 3,9%. Ετήσιο έλλειμμα ανέβηκε στο 4% ενώ πέρσι ήμασταν στο 3,3% και φέτος θα ε, ξαναπέσουμε κάτω από το 3%. Επομένως θα εκπληρώσουμε αυτό το κριτήριο της ηθίκης του Μάστριχτ. Το πρόγραμμα σταθερότητες ετησίως επηρεάζει αρνητικά την οικονομία κατά μισή μονάδα του ΑΕΠ ετησίως και θα έχουμε πρόγραμμα σταθερότητας μέχρι το 2016. Τώρα ως προς το διαρθρωτικό έλλειμμα, ένα γερμανικό οικονομικό ίδρυμα υπολόγισε 62 διαφορετικά διαρθρωτικά ελλείμματα για τη Γερμανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξεπλάγει διότι η γερμανική κυβέρνηση ανακάλυψε και ένα 63ο ε, διαρθρωτικό έλλειμμα το οποίο δεν είχαν ανακαλύψει αυτοί από αυτό το γερμανικό ερευνητικό ίδρυμα το οποίο ε, ήταν υπόλογο ε, για δύο μονάδες του ΑΕΠ. Επομένως το ερώτημα σε σχέση με τα διαρθρωτικά ελλείμματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και προς το παρόν καλό, καλό είναι να μην το πάρουμε στα σοβαρά. Δηλαδή ό,τι και να λέει κάποιος για το συγκεκριμένο διαρθρωτικό έλλειμμα μιας χώρας δεν θα πρέπει να ε, παίρνετε πολύ στα σοβαρά. Ε, τώρα, ως προς το φόρο επί των χρηματιστηριακών ε, συναλλαγών, ξέρετε, αν αγοράσετε ένα λίτρο γάλα θα πληρώσετε 10% ΦΠΑ στη δική μου χώρα αν αγοράσετε κάτι άλλο θα πληρώσετε 20% φόρα. Αλλά αν αγοράσετε κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή σας, όπως είναι μια μετοχή ή μια οψιόν, ένα δικαίωμα προαίρεσης, δεν θα πληρώσετε καθόλου φόρο. Κανείς δεν μου έχει εξηγήσει τι είναι τόσο το, ποιο είναι το φοβερό με το γάλα που πρέπει να φορολογείται και ποιο είναι το τόσο ε, εκπληκτικό με τη μετοχή το δικαίωμα περιόρισης που δεν πρέπει να φορολογείται. Αν δεν είναι βεβαίως η φόρο αποφυγή. Καλό είναι να έχουμε διαφορετικούς φόρους και να υπάρχει ανταγωνισμός για το ποιος θα έχει χαμηλότερη φορολογία. Αυτό είναι καλό, συμφωνώ. Για ποιους όμως θα έχουμε χαμηλότερη φορολογία. Μόνο για αυτούς που είναι στο πάνω μέρος, στην κορυφή της ιεραρχίας, το 1% και μάλιστα αν θέλετε και το 1% των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν λιγότερο από 1% του λαού. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό μόνο για τους εξαιρετικά ε, πλούσιους ή είμαστε εδώ για να καταστήσουμε σαφές ότι και αυτοί πρέπει να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, μου μένουν δύο λεπτά για τις υπόλοιπες 300 ερωτήσεις. Καταρχάς, Πολλοί αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην ολοκλήρωση της νέας αγοράς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μία σειρά 20 μέτρων έχουν υιοθετηθεί και στη δική μου επιτροπή για το Ταμείο Κοινωνικών Επενδύσεων, ε, για τα κεφάλαια πάρα πολλά μέτρα για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ε, τα οποία θα εξεταστούν και θα εφαρμοστούν βάσει της διαδικασίας fast track. Και θέλω να τονίσω ότι και στην εξάδα των μέτρων και στη μήνυ συνθήκη και στο ε, Pact Plus ε, αναφέρονται, στο Plus Pact αναφέρονται όλα αυτά. Προγραμματίζεται τα ομόλογα έργου με μόχλευση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα δρομολογήσουμε ε, και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει το ευθύνη ε, που του αναλογεί προσπαθώντας να προωθήσει φόρο επί των χρηματιστηριακών ε, συναλλαγών και όχι επί των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών και ίσως σε βάθος χρόνου τελικά οριμάσει αυτή η ιδέα περισσότερο και καταστεί εφικτό να ενσωματωθούν και οι δραστηριότητες οι χρηματιστηριακές και όχι μόνο οι συναλλαγές. Ορισμένοι είπαν ότι δεν έχουμε αρκετούς κανονισμούς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εγώ έχω 29 μέτρα αυτή τη στιγμή τα οποία χειρίζαμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συντονίσουμε τις ε, ε, καθευτήρες γραμμές για τις μακροπιστώσεις, ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, π.χ. το Ιρλανδικό πρόβλημα, να εντοπίζονται καιρός φούσκες, οι ανισορροπίες στα συστήματα. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν εξαιρετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδιοργανωθεί ο οικονομικός διάλογος, να τονίσουμε ότι και το Βέλγιο και η Ουγγαρία ε, συμφώνησαν να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής μας. Δεν είναι κλίση υποχρεωτικής παράστασης. Τους δίνουμε μια ευκαιρία να εξηγήσουν. Εάν θέλουν την αξιοποιούν, δεν είναι υποχρεωτικό. Ε, επιλέγουν γιατί θέλουν να ε, εισπνεύσουν το οξυγόνο της δημοσιότητας, εμφανιζόμενοι δημοσίως ενώπιον της Επιτροπής ή δεν επιθυμούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την κοινωνία, αν θέλετε, από τη στιγμή που όλοι ε, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, όλοι πληρώνουμε το τίμημα. Άρα είναι αναγκαίο να έχουμε συλλογική στήριξη από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας και όχι μόνο από ένα κράτος μέλος. Και η τελευταία παρατήρηση μου έχει να κάνει με αυτό που ο Φιλανδός συνάδελφος για τα επιτόκια. Καταλαβαίνω το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου το οποίο προβάλλεται. Νομίζω όμως ότι όσοι συμβάλλουν στα προγράμματα αυτά, όσοι υφίστανται τα προγράμματα αυτά, ήδη πληρώνουν ψηλό τίμημα για παρελθόντα αμαρτήματα και δεν θα πρέπει να υφίστανται αυτή τη βύση των απίστευτα υψηλών επιτοκίων. Στην Ελλάδα για να φτάσει στο 120 του ΑΕΠ ε, το χρέος χρειάζονται άλλα 8 χρόνια αν τα καταφέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι το τίμημα είναι υψηλό. Μπορούμε με τα ευρωμόλογα να έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει πειθαρχία αλλά και να ε, δοθεί ευκαιρία για ένα δεύτερο γύρο ε, σε βραχυπρόθεσμη βάση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γύρω από την ε, νομική έννοια του ηθικού κινδύνου. Μία πολύ σωστή παρατήρηση που έγινε στη συζήτηση κατά την άποψή μου είναι η εξής. Χρειαζόμαστε πράγματι περισσότερη Ευρώπη, αλλά ε, εν ευθέτω χρόνο, τη, στη σωστή χρονική στιγμή. Και αυτό έχει άμεση σχέση με πολλά από τα μέτρα που εξετάζουμε και που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Ε, πλησιάζει 7 η ώρα. Να σας πω ότι στο εστιατόριο ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρατεθεί δείπνο και αύριο θα συναντηθούμε ξανά στις 9 σε αυτήν εδώ την αίθουσα και θα μιλήσουμε για τη συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ποια συνέχεια θα δοθεί. Άρα θα αποτελέσει αυτό συνέχιση των συζητήσεων που ε, είχαμε σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. If, if you want to hang αν θέλετε να ε, παραμείνετε εδώ κοντά για να σας δείξουν η βοηθή που είναι το εστιατόριο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε, ε, ε, γρήγορα θα έρθει κάποιος να σας βοηθήσει.